Good morning Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αναφορών στη σημερινή μας συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε και εσείς αναφερόμενοι και αναφερόμενες καθώς και όλες και όλοι όσοι παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Καθίστε και όποιοι επιθυμείτε θα λάβετε το λόγο. Το θέμα υπαριθμών 2 είναι έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Το 53β έχει καταργηθεί. Λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες και δεν κλείνει η αναφορά. Αν δεν υπάρχουν ε, άλλες ενστάσεις, τότε εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Στο υπαριθμόν 3 εγκρίνουμε τα πρακτικά της ε, 18, η συγγνώμη, 19 Απριλίου του 2016. Δεν έχω ανακοινώσεις της Προέδρου. Αυτά θα τα πούμε μετά το μεσημεριανό γεύμα. Θα σας εξηγήσω τότε και τι έγινε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Δυστυχώς δεν θα είμαι σήμερα. Ε, πρέπει να επιστρέψω στη Σουηδία ταχύτατα, διότι ο γιος μου αποφυτά αύριο. Όμως η Αντιπρόεδρος θα είναι εδώ και Είμαι βεβαία ότι θα διευθύνει με θαυμάσιο τρόπο την συζήτηση. Ε, στα διάφορα δεν έχω τίποτε, ούτε έχει ζητήσει κανείς τον λόγο για ε, κάποιο θέμα στα διάφορα. Ας έλθουμε τώρα στην αναφορά 0446 του Χάρι Σίνφλερ. Έχω ζητήσει το λόγο για ένα λεπτό, ε, λέει ένας ευρωβουλευτής. Ναι, ναι, η πρόεδρος. Για την υπαριθμόν 51, έτσι δεν είναι. Πρόκειται για αποζημιώσεις. Γνωρίζω ότι θα συζητηθεί το Σεπτέμβριο το θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να πω λίγα λόγια και έχω και μια ερώτηση. Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή σας αποφάσισε να στείλει επιστολές στην ε, γερμανική κυβέρνηση και στην ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε λάβει απάντηση από τις αρμόδιες αρχές και ποιο είναι το περιεχόμενο της απάντησης αυτής. Και ένα ακόμα, εκ μέρου των αναφερομένων. Ζητούν από, μάγνια η στάση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων είναι απαράδεκτη και προκλητική. Λέει δηλαδή ότι το θέμα είναι διμερές μεταξύ των δύο χωρών και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρέμβει. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει σε πολλές διμερείς διαφορές, ακόμα και εσωτερικέ διαφορές απανταχού του κόσμου. Ακόμα και δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Λέει ο κύριος Ζαϊρανόπουλος. Ε, πρέπει να τεθεί το θέμα ώστε να μπορέσει να συζητηθεί και περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την μεταπολεμική διεθνή συνθήκη για τις πολεμικές αποζημιώσεις της Γερμανίας επί, της, επί, επί του οποίου κειμένου βασίζεται το ελληνικό δικαίωμα για επανορθώσεις. Το σέβεται το κείμενο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. επί του θέματος το οποίο τέθηκε. Θέλω να πω ότι η αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, η οποία τέθηκε υπόψη μας, μετά από συζήτηση και εισήγηση δική μου, κρίθηκε παραδεκτή. Και μετά από αυτό έφυγαν επιστολές στην Κομισιόν, στην, Επιτροπή, στην ελληνική κυβέρνηση και προς την γερμανική κυβέρνηση. Ε, Εν συνεχεία είχαμε την άποψη της Κομισιόν ότι δήθεν η αναφορά δεν είναι παραδεκτή, μάλλον ότι η αναφορά δήθεν δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντικείμενο και ότι θα πρέπει να απορριφθεί. Η θέση αυτή έχει αντικρουστεί αρκετές φορές από την πλευρά τη δική μας, διότι το θέμα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση Ούτως ή άλλως η Ελλάδα και η Γερμανία δεν έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης. Επομένως είναι ένα θέμα σοβαρό το οποίο ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή μας. Είναι ένα θέμα που αφορά τους αναφέροντες διότι είναι πολλοί από αυτούς εκφράζουν τους συγγενείς των θυμάτων χιλιάδων πολιτών Ελλήνων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Εξηγήσαμε ότι είναι εντός της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πέραν των άλλων αφορά και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που επηρεάζει τα ζητήματα της ε, δημοσιονομικής λειτουργίας της Ένωσης ε, και τον ελληνικό προϋπολογισμό. Διότι εγγραφόμενες οι αποζημιώσεις στον προπολογισμό της Ελλάδος θα μετατρέψουν τον προϋπολογισμό σε πλεονασματικό. Επομένως αφορά την ίδια τη λειτουργία και της Ευρωζώνης. Αυτά όλα τα επιχειρήματα τέθηκαν υπόψη και ε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ε, επειδή την προηγούμενη Παρασκευή από πλευράς μας ασκήσαμε γραπτές αντιρρήσεις επί της προτάσεως της Γραμματείας της Επιτροπής να κλείσει η υπόθεση, θεωρούμε σημαντικό το ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Θα φέρουμε, I'm going to finish in 20 seconds. Θα φέρουμε τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται επιπλέον για να πιστεί η Επιτροπή ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να προχωρήσει και στο έγγραφο που έχω κάνει κυρία Πρόεδρε προς την Επιτροπή σας ζητώ να στείλετε έγγραφο στην ελληνική και γερμανική κυβέρνηση να παρουσιάσουν εγγράφος τις απόψεις τους για το θέμα αυτό. Επομένως, οψόμεθα στις 8 Σεπτεμβρίου για το ζήτημα αυτό, παρότι βεβαίως οι αναφέροντες έχουν διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της Γραμματείας να κλείσει την υπόθεση αυτή. Θεωρώ σημαντική την απόφασή μας ως συντονιστές ότι διατηρούμε ανοιχτή την υπόθεση αυτή μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου και θα είμαστε εδώ για να θέσουμε αναλυτικά όλα τα επιχειρήματα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Okay. So... Η πρόεδρος. 51. Ο κύριος Μαριάς ζήτησε ήδη να εξαιρεθεί του καταλόγου. Εδώ ε, ισχύει ο κανόνας των δύο μηνών. Άρα μετά το καλοκαίρι θα το ξανασυζητήσουμε. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη ωστόσο σήμερα. Αλλά δεν έχει κλείσει. Και σε ό,τι αφορά τις επιστολές, στάλθηκαν στην ε, μόνιμη αντιπροσωπεία για ενημέρωση. Αυτό είναι. Νομίζω ότι με αυτά πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση αυτή δεν είναι στην ημερησία διάταξη σήμερα. Εμεί συζητούμε τα όσα βρίσκονται στην ημερησία διάταξη σήμερα, δηλαδή το 446, την αναφορά 446-2007. Αν θέλετε παραμένετε, αν θέλετε επανέρχεστε όταν θα ε, τεθεί το θέμα σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ζακλίν Κοτρέλ και Ζακλίν Μακλένεν που είναι εδώ για την αναφορά 557. Έχετε το λόγο. Good morning. Έχω μεγάλο σεβασμό για την Επιτροπή Αναφορών. Έχω δει και τις παρεμβάσεις των βουλευτών και της γραμματείας. Δυστυχώς δεν είναι θετικά τα ε, αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το δικαίωμά μου να ψηφίσω. Έρχομαι στην αναφορά του κ. Σίντλερ, δηλαδή τη στέρηση του δικαίωματο ψήφου Βρετανού υπηκόου, που δηλαδή στερείται το δικαίωμα του εκλέγην εάν έχει διαμείνει στο εξωτερικό επί 15 έτη. Αποκλείεται λοιπόν από, την, ε, από το δικαίωμα ψήφου. Και αυτό αφορά μεγάλους αριθμούς Βρετανών πλησιάζουμε σε λίγες εβδομάδες στο Βρετανικό δημοψήφισμα. Εκεί θα έπρεπε να ακουστεί η φωνή όλων των Βρετανών υπηκών. Εγώ είμαι μία από τις Βρετανίδες υπηκός. Όμως η ε, Βρετανική Βουλή ψήφισε νόμο που περιλαμβάνει τον κανόνα των 15 ετών και δεν έχω το δικαίωμα πλέον να ψηφίσω. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματά μας διαμένοντας στην Αλοδαπή, εκτός δηλαδή Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό όμως μας στερεί το δικαίωμα του εκλέγην. πρόκειται για παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας και πρέπει να ανατραπεί ο κανόνας αυτός. Έχουν προειδοποιηθεί ήδη τα θεσμικά όργανα και πρόκειται για μια μεγάλη αδικία. Και η Επιτροπή Αναφορών και η Κομισιόν έχουν συμφωνήσει ότι χρειάζεται να ληφθεί δράση. Στην ανακοίνωσή της του 2014 η Κομισιόν προτείνει σχετικά μέτρα στις χώρες μέλη. Επίσης η Βρετανική Επιτροπή Αναφορών απήντησε σε επιστολή σας είπε ότι θα ζητήσει από την ε, Βρετανική κυβέρνηση να υποβάλει ε, πρόταση νόμου που να αποκαθιστά το δικαίωμα των όσων Βρετανών υπηκών ζουν στην Ολοδαπή επί 15 χρόνια και μετά. Όμως ακόμα δεν έχει γίνει αυτό και δεν προλαβαίνει να γίνει μέχρι το δημοψήφισμα. Όσοι εξημών υφιστάμεθα στέρηση των δικαιωμάτων μας, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να διατηρήσει τα πλήρη μας δικαιώματα ως Βρετανών υπηκών. Πρόκειται για στέρηση του δικαιώματος ε, ψήφου, ε, του εκλογικού δικαιώματος δηλαδή, εκατομμυρίων Βρετανών πολιτών που διαμένουν στην Αλοδαπή. Παρόλε τις προσπάθειές μας δεν έχει αναλυφθεί καμιά δράση. Είμαι εκλεγμένη δημοτική ε, σύμβουλος στην Ισπανία. Η κόρη μου που θα γίνει 30 ετών φέτος δεν μπόρεσε να ψηφίσει ποτέ μέχρι τώρα, ούτε στην Ισπανία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήμερα υφίσταται την μομφή ότι είναι αντιδημοκρατική, είναι πιο ζωτική σημασία από ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσουν ταχαίω ώστε να διατηρηθούν τα δικαιώματα όλων αυτών των προσώπων το, στις ε, συστάσεις του 2014 είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το δικαίωμα του εκλέγην είναι βασικό, θεμελιώδες δικαίωμα ε, του πολίτου. Είναι δυνατόν να υπάρξουν λύσεις. Υπάρχουν επιχειρήματα που έχουν, ε, που έχουν υποβληθεί με νομικά έγγραφα και πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Ο συνεχιζόμενος πολιτικός διάλογος θα επιτρέψει στην Επιτροπή Αναφορών, στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να εξετάζουν το ζήτημα αυτό για να μπορούν οι Βρετανοί υπήκοοι να ψηφίζουν στην χώρα διαμονής τους, όπως είχε περιληφθεί ως πρόταση και στην ανακοίνωση του 2014. Θα παρακαλέσω, θα ρωτήσω μάλλον τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη τα διαβήματα αυτά από τις χώρες Μπέρι, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φροντίζει ώστε να εφαρμοστούν οι συστάσεις της και να επεκταθεί το δικαίωμα ψήφου των Βρετανών υπηκών στις χώρες διαμονής τους. Είμαι μια πεπισμένη Ευρωπαία και εξακολουθώ να πιστεύω ότι με, και, την, σε ένα μήνα ακόμη θα είμαι ε, Ευρωπαία πολίτης. Όμως χρειάζεται ανάπτυξη δράσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ποτέ πια ε, ένας, Βρετα... ένας ε, Ευρωπαίος πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να χάσει την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη επειδή δεν θα μπορεί να ψηφίσει ή επειδή η χώρα του θα αποχωρήσει. Πρέπει να ε, ταχθούμε υπέρ όλων των δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών να μπορούν δηλαδή να ψηφίσουν στη χώρα που έχουν επιλέξει ως πατρίδα τους. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση για να συνεχιστεί ο αγώνα αυτό για την εξασφάλιση των δημοκρατικών μα δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε και θα διατηρήσετε ανοιχτή την αναφορά αυτή, ώστε να μπορέσει να επιληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρο. Ορίστε, συνεχίστε, αλλά ε, κάπω πιο σύντομα αν γίνεται. Διότι ε, για διαφόρου λόγου έχουμε περιορισμένο χρόνο. Δεν έχει μικρόφωνο. αξιότιμοι ευρωβουλευτές και αξιότιμες ευρωβουλευτές. Λέγομαι Τζάκλιν Μακλέναν, εκπροσωπώ τον αναφερόμενο RC για την αναφορά του με θέμα ότι το Ενωμένο Βασίλειο δεν επιτρέπεται να αποκλείσει όσους Βρετανούς πολίτες βρίσκονται ε, στην Αλοταπή για παραπάνω από 15 χρόνια από το να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα, διότι το αποτέλεσμά του μπορεί να έχει σοβαρέτατες συνέπειες στην κατάστασή τους. Ε, βεβαίως το δημοψήφισμα αυτό που εννοεί και είπε και η προηγουμένη ε, ομιλήτρια, είναι το ε, δημοσίευμα της 23ης Ιουνίου που ε, ενδέχεται να οδηγήσει έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ένωση. Εγκρίθηκε νόμος στο Δεκέμβριο του 2015 από τη Μεγάλη Βρετανία και περιλαμβάνει τον κανόνα των 15 ετών που απαγορεύει στους Βρετανούς που διαμένουν 15 χρόνια και περισσότερα εκτός Μεγάλης Βρετανίας από το να συμμετέχουν είτε σε γενικές εκλογές είτε και σε δημοψηφίσματα. Έτσι λοιπόν ο αναφερόμενος RC που είναι Βρετανός υπήκος και διαμένει στην Ιταλία από το 1993 αλλά και εγώ που είμαι Βρετανίδα υπήκος και ζω και εργάζομαι στο Βέλγιο από το 1987 και οι δυο έχουμε χάσει το δικαίωμά μας να ψηφίζουμε και το δικαίωμά μας αυτό ψήφου, δηλαδή η συμμετοχή στις εκλογές στην πατρίδα μας είναι βασικό θεμελιώδες δικαίωμα. Και για τον αναφερόμενο Αρσί, αλλά και για μένα, θεωρούμε ότι αυτό είναι παράνομο και αντιδημοκρατικό. Θίγονται δε περίπου 2 εκατομμύρια Βρετανοί πολίτες που δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα. Η άποψή μου είναι, δεν είναι καμιά επαναστατική άποψη, υποστηρίζεται και από την ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση και όπως είπε και η άλλη συναναφερομένη, η Βρετανική κυβέρνηση ίδια δέχθηκε ότι πρέπει να αλλάξει ο κανόνας αυτός. Είπε όμως ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό πριν από την εξαγωγή του δημοψηφίσματος. Αυτή ήταν η θέση της Βρετανικής κυβερνήσεως και είναι στην πραγματικότητα μια ντροπιαστική για την ίδια θέση. Μαζί με τον κύριο Χάρι Σίντλερ, εγώ κατέθεσα αναφορά για το Βρετανικό δημοψήφισμα και προέβαλα το επιχείρημα ότι ο σχετικός, βρετανικό ε, Βρετανικός νόμος είναι παράνομος διότι έρχεται σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο το οποίο εξασφαλίζει την ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης η ίδια δηλαδή η συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είπα μάλιστα ότι ο κανόνα αυτό αποτρέπει του πολίτε από το να χρησιμοποιούν τα δικαιώματά του που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Και ότι είναι και συνταγματικό. Τις τελευταίες εβδομάδες στραφήκαμε στα δικαστήρια, σε τρία δικαστήρια τριών διαφορετικών βαθμίδων στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώ απορρίφθηκαν τα επιχειρήματά μα από τι τρει αυτέ βαθμίδε. Εμεί επιχειρηματολογήσαμε ότι εάν χάσουμε, εάν δηλαδή τελικώ το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ηνωμένη Ευρώπη, εμεί δεν θα είμαστε πλέον ω Βρετανίδε υπήκοοι, δεν θα είμαστε ε, Ευρωπαίοι πολίτες. Θα καταλήξω να είμαι γκάσταρμπάιτερ στο Βέλγιο. Το αποτέλεσμα θα έχει βαθύτατες επιπτώσεις σε ανθρώπους όπως ε, εγώ. Πολύ περισσότερο από τους Βρετανούς πολίτες που είναι εγκατεστημένοι στο, ε, Μεγάλο Βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγγνώμη. Το δικαστήριο όμως δεν συμφώνησε. Εμείς έχουμε το άρθρο 50 της, ε, σε, νέο, σε, νέα, σε νέο, σχέδιο συνθήκης θα υπάρχει κανόνας, υποτίθεται, ο οποίος επιτρέπει σε χώρα μέλος να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εμείς θέλουμε να μπορούμε να ψηφίζουμε σε δημοψηφίσματα τόσο μεγάλης εμβέλειας. Η ηρωνία και η ασυνέπεια της καταστάσεως αυτής έγινε στο εξής στερούνται οι Βρετανοί υπήκοοι θεμελιώδη δικαιώματά του, Μόνο και μόνο διότι άσκησαν θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία του έχουν παραχωρηθεί από την συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την ελευθερία εγκατάστασή του. Απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Χάρη Σίντερ με επιστολή και είπε ότι η σύσταση που εγκρίθηκε και προσκαλεί τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες τους θα συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα συμμετοχή στις εκλογές και ότι αυτό αποτελεί μια ισορροπημένη προσέγγιση. Για μένα αυτό δεν είναι επαρκέ. Εγώ ζητώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που αναγνωρίζουν ότι η πλήρη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα αποτελεί την πεμπτουσία της ε, ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Τα θεσμικά όργανα οφείλουν να το αναγνωρίσουν αυτό και έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ώστε τα δικαιώματα των πολιτών αυτών να διατηρούνται, να γίνονται σεβαστά σε όλε τι χώρε μέλη. Κάτι το οποίο δεν έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Χάρη Σίνερ και εγώ αναγκαστήκαμε να στραφούμε στα Βρετανικά δικαστήρια. Όπου, όπω σα είπα, τα επιχειρήματά μα απορρίφθηκαν. Τώρα στρεφόμαστε στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι σα ξαναείπα ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει δυσμενώ 2 εκατομμύρια Βρετανούς πολίτες. Σας παρακαλώ να αποκαταστήσετε το δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ για την ε, συνεισφορά σας, λέει Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν όντω θεωρεί πω είναι πολύ σοβαρό, να, πολύ σημαντικό να προωθηθεί η πλήρη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι και ο λόγος που το 2014 αναφέρθηκε από, και από τους αναφέροντες υιοθετήθηκε η σύσταση για το δικαίωμα συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης στα, κράτος, στα κράτη-μέλη για τους πολίτες που χρησιμοποιούν την τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ένωση. Ωστόσο, πρόκειται για σύσταση και όχι για δεσμευτικό ε, μέσο. Όμως αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη, στην Κομισιόν να καλέσει τα κράτη-μέλη μεταξύ αυτών και του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκολύνουν ε, τους ε, υπηκόστους που έχουν χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας να διατηρήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές εκλογές εφόσον επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την πολιτική ζωή της χώρας. Η Κομισιόν παρακολουθεί τις συζητήσεις και τις εξελίξεις ε, σε αυτό το θέμα και υπάρχει συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, επεκτείνει την δυνατότητα αυτή για τους, για τους ε, Βρετανούς πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, να μπορούν δηλαδή να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές και επίσης ε, αυτό ισχύει για τους κατοίκους που έχουν διαμείνει 15 χρόνια στην Αλοδαπή να μπορούν να ψηφίσουν και στις Βρετανικές εκλογές. Ωστόσο, η Κομισιόν δεν έχει τις δυνατότητες να παρέμβει στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις εκλογές. Η συνθήκη θα δίνει ε, δικαιώματα. Είναι το άρθρο 22β, δεν κάνω λάθος. Ε, το δικαίωμα να είναι κανείς υποψήφιος και να συμμετέχει στις εκλογές υπό τις ίδιους όρους όπως η υπηκόη του εν λόγω κράτους. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει γενικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να ψηφίζουν σε εθνικά δημοψηφίσματα. Ε, η διοργάνωση δημοψηφισμάτων εμπίπτει απολύτως στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Υπό λοιπόν των όσων μόλις σας είπα, δεν είμαστε σε θέση η Κομισιόν τουλάχιστον, να διαπιστώσουμε παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε αυτές τις υποθέσεις και λυπούμεθα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Και τώρα οι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Πρώτη είναι η Τζούντι Κέρτεν Darling. Πριν να σου δώσω όμω το λόγο. Εξ ονόματο των συναδέλφων και η μου τη ιδία, να σε συγχαρώ για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι τα γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά τα γενέθλια δεν έχουν και πολύ σημαντικά όταν έχουμε εδώ δημοψηφίσματα που αφορούν το μέλλον της χώρας. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τους ε, αναφέροντες που είναι σήμερα εδώ και που ε, παρουσιάζουν τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους στην Επιτροπή. Εδώ αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ καιρό και είναι κρίμα που τρεις εβδομάδες μόλις πριν από το ευρωπαϊκό δημοψήφισμα επανέρχεται. Ε, μπορεί να κάνουμε ένα σωρό ωραίες δηλώσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι, όπως είπαν και οι δύο ε, αναφέρουσες, ότι τώρα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις προθεσμίες όσον αφορά την γραφή ε, στο Μητρώα για τους Βρετανούς ε, κατοίκους. Αυτό η προθεσμία ε, τελειώνει σε πέντε μέρες μόλις, οπότε πραγματικά είμαστε στην τελευταία ευθεία, στην τελική ευθεία πριν το δημοψήφισμα. Τώρα όμως όσον αφορά την επέκταση της δυνατότητας σε ευρύτερε ομάδες, και ως πολιτικός του Εργατικού Κόμματος θα σας πω ότι το Εργατικό Κόμμα δεν έλαβε θέση υπέρ της ε, κατάργησης του κανόνα των 15 ετών. Η βασική μας προτεραιότητα σε σχέση με αυτό το δημοψήφισμα ήταν να εξασφαλίσουμε πως οι νέοι που θα επηρεαστούν πολύ λόγω των αποτελεσμάτων θα συμμετέχουν. χρόνια επιτρέπεται να ψηφίσουν στη Σκωτία για το αν θέλουν να μείνουν ε, στην Ένωση ή όχι ε, για το αν θέλουν μάλλον να μείνουν εντό του Ηνωμένου Βασιλείου ή όχι. Υπάρχουν τρει ομάδε που επηρεάζονται περισσότερο και ωστόσο δεν έχουν φωνή. Είναι οι νέοι που θα επηρεαστούν στη διάρκεια ολόκληρη τη ζωή του από αυτή την απόφαση για το αν θα μείνουμε ή αν θα φύγουμε. Η δεύτερη ομάδα είναι οι Ευρωπαίοι που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί λέμε συχνά για Ευρωπαίους ε, μετανάστες και ε, Βρετανούς εκπατρισμένους Άρα λοιπόν Ευρωπαίοι εκπατρισμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν ακόμα και αν μένουν εκεί, πληρώνουν τους φόρους τους και συμβάλλουν στην, ευρωπαϊκή, ε, στην, συγγνώμη, στην Βρετανική οικονομία. Και οι άνθρωποι που ζουν εκτός Βρετανίας για πάνω από 15 χρόνια δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Είναι αυτό τραγική ηρωνία. Δύο εκατομμύρια κόσμος είναι που πραγματικά αντιπροσωπεύουν τη Βρετανία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στα όργανα λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής. Εργάζονται προς το συμφέρον της χώρας μας στο εξωτερικό. Είναι και άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να ε, εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Και λυπάμαι πολύ που οι τρεις αυτές ομάδες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα. Τούτου λεχθέντος δεν είμαστε η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Η Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Ουγγαρία, Μάλτα επηρεάζονται από περιορισμούς για τους υπηκόους τους που ζουν αλλού. Και είναι ευρύτερο το ζήτημα αυτό. Και αυτό είναι και η ουσία ε, για αυτή την Επιτροπή Αναφορών. Ελπίζω ότι θα είμαι μέλος της Επιτροπής Αναφορών μετά από τις 23 Ιουνίου, γιατί εμείς είμαστε υπέρ του να παραμείνουμε στην Ένωση και άρα να μπορέσουμε να παρατείνουμε, να επεκτείνουμε μάλλον αυτά τα ωφέλη για τον κόσμο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί η ευρωπαϊκή λύση. Πολλά έχουν υποθεί για, από τις αναφέρουσες και την Κομισιόν για τις δράσεις που ήδη έχουν γίνει από τη Βιβια Ρέντινγκ ως Επίτροπο είτε από τον Φρέντς Τίμερμανς. Κρίσιμο ε, η παρατήρηση είναι ότι εφόσον υπάρχει ελευθερία κυκλοφορία, αυτό θα πρέπει να καταλήξει στην ε, στέρηση του δικαιώματος ψήφου εντός της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να υπάρξει αλλαγή. Το, 1900, το 2015 ο Επίτροπος Σίμερμαν ήρθε στην Επιτροπή Αναφορών και απάντησε ερωτήσεις δικές μας για τα δικαιώματα ψήφου και την ε, υπηκότητα και δεσμεύτηκε ότι θα ανελάμβανε τον ρόλο του ενδιάμεσου με τα κράτη-μέλη εκεί όπου τα δικαιώματα ψήφου δεν ε, ήταν ε, πολύ εκτεταμένα και θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν τι έχει γίνει εντωμεταξύ. Έχει γίνει κάτι. Έχουν γίνει διαβήματα προς την Βρετανική κυβέρνηση και τις υπόλοιπες κυβερνήσεις ε, που κρατούν την ίδια στάση. Η Κομισιόν στην ουσία είναι της άποψης πως αυτά είναι τα πράγματα, έτσι είναι τα πράγματα και δεν, να γίνει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Γιατί φοβούμαι από την απάντηση που άκουσα από την Κομισιόν ότι αυτή τη στάση κράτησαν. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτό είναι, ε, αυτό είναι το βασικό ερώτημα επιτάπητος ε, σήμερα. Ξέρουμε ότι όλα αυτά έχουν περιγραφεί και στις συστάσεις. Τι άλλες ε, ενέργειες μπορούμε εμείς να κάνουμε και εμείς ως Επιτροπή Αναφορών μπορούμε να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις να έρθουν και να ξεκινήσουν διάλογο με το Ευρωκοινοβούλιο. Εάν η Κομισιόν δεν μπορεί να, να κάνει κάτι, μπορεί να κάνει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Άντζελα. Ευχαριστώ κάθε μέρα. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ τις αναφέρουσες καταλήγει σε ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η κατάσταση που περιγράψανε δεν είναι μοναδική περίπτωση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μου το ζουν οι εκατοντάδε χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από την Ισπανία για να δουλέψουν αλλού, είτε προσωρινά είτε μονίμως. Για να καταλαβαίνουμε όλοι περί τίνος πρόκειται, στις εκλογές του 2014 τις περιφερειακές και τις τοπικές μόνο το 3,2% αυτών που κατοικούν στο εξωτερικό ψήφισαν και στη, το 2014 στις ευρωεκλογές επίσης πάρα πολύ λίγοι. Οπότε οι χιλιάδες άνθρωποι που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν γιατί περιλαμβάνονται στους ε, καταλόγους μόνο το 0,6% το έκανε. Και δεν είναι επειδή δεν ενδιαφέρονται, αλλά για πολλούς λόγους. Γιατί υπάρχουν περιορισμένες προθεσμίες, υπάρχουν γραφειοκρατικά κολλήματα κλπ. κλπ. Είναι μια κατάσταση λοιπόν άδικη, η οποία πλήττει και το δικαίωμα ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήτη και την αρχή της δημοκρατίας, της μη διάκρισης και το δικαίωμα της ισότητας απέναντι στον νόμο που περιλαμβάνεται και στη Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων και στις συνθήκες μας. Συνεπώς, φυσικά και πρέπει να ζητήσουμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή, μαζί και με άλλες αντίστοιχες αναφορές από άλλες χώρες, όπως και η δικιά μου, ε, να μπουν μαζί σε μια ομάδα, να τη συζητήσουμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μη τι άλλο, να κάνει μια αξιολόγηση τη σύσταση του 2014 που ζητούσε μέτρα προκειμένου οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα τη ελεύθερη κυκλοφορία του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να απαντήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώρε ακολούθησαν τι συστάσει να υπάρξει μια έκθεση για τα αποτελέσματα των συστάσεων αυτών και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, όπως επίσης και τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάψει αυτή η υπερθωριοποίηση, αυτή η στέρηση ενός τόσο θεμελιωδούς ε, δικαιώματος όπως είναι εκείνο της, ε, του εκλέγην και εκλέγεστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Σολεδάδ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα. Η αρχή της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας βασίζεται στο θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης σε όποια χώρα της επιθυμεί κανείς. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα που συνοδεύουν αυτό το δικαίωμα, αλλά αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει ένα κενό όμως, ένα κενό για το πού ψηφίζει κανείς, πού έχει το δικαίωμα να σκίσει αυτό ακριβώς το δικαίωμα ψήφου του κανείς. Η μη ρύθμιση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, πλήττει το δικαίωμα αυτό στις εθνικές εκλογές. Έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα, ακούσαμε ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες, υπάρχει το θέμα με την Βρετανική υπηκότητα. Τόσο για αυτούς που ζουν μέσα όσο και εκτός του Ενωμένου Βασιλείου όπου η ερμηνεία αυτή της επικότητας γίνεται περιοριστικά, αποκλείονται δηλαδή κάποιοι. Οπότε πιστεύω ότι το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές πρέπει να συνδέεται με την υπηκότητα, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση πρέπει να υπάρχει βέβαια συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρξει αλλαγή και το δικαίωμα δίνεται για να ψηφίσει κανείς εκεί που κατοικεί. Οπότε, το πρόβλημα είναι πρόβλημα βρετανικής νομοθεσίας. Ε, το Κοινοβούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια αποφασίζει βάσει της νομοθεσίας που ισχύει εκεί. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αφού πλήττεται ένα θεμελιώδες δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών εξαιτίας της εθνικής αυτής νομοθεσίας. Να γίνει μια σοβαρή ελεύθερη συζήτηση για αυτό το βασικό δικαίωμα που είναι το δικαίωμα της ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που πλήττεται σε κάποιες χώρες. Οπότε, απλώς ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Σε λίγε μέρε θα έχουμε δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο με το οποίο θα αποφασιστεί κατά πόσο θα μείνει ή θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η χώρα. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, πολύ ευαίσθητο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με του Βρετανού πολίτε και αργότερα στην Επιτροπή μα να συζητάμε αυτό το θέμα, γιατί εννοείται ότι ανήκουν στην Ευρώπη και πρέπει να μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα, ευχαριστούμε. Πάλι. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σλοβακικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμείς χαιρόμαστε όταν βλέπουμε να αγωνίζονται οι πολίτες υπέρ των δικαιωμάτων τους. Πρόκειται για βασική αρχή της δημοκρατίας. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία αυτή. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα και γι' αυτό χαίρομαι που το συζητούμε εδώ. Και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο σχετικά, ώστε να πείσουμε τις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν περιοριστικά το ζήτημα αυτό, να προσαρμόσουν τα δικαιικά του συστήματα και μάλιστα να τα προσαρμόσουν θετικά. Σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη κατάσταση, θα πω το εξής Χαίρομαι που η κυβέρνηση του Ενωμένου Βασιλείου εκφράζει την επιθυμία να τροποποιήσει το σχετικό νόμο. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για το πότε, το πώς και το εάν θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ε, αναφερομένων. Ίσως είναι δυνατόν να στραφούμε προς τα ε, αρμόδια θεσμικά όργανα της Βρετανική ε, για να μας παράσχουν τις σχετικές πληροφορίε. Πάντω, με μεγάλη μου λύπη θέλω να τονίσω ότι προφανώς η λύση αυτή δεν θα προλάβει να ισχύσει πριν από το δημοψήφισμα τη 23 η Ιουνίου. Και στο όνομα του Λαϊκού Κόμματος εύχομαι κάθε επιτυχία στις και στου πολίτες που επιθυμούν η χώρα του να παραμείνει στην Ένωση. Ευχαριστώ. Η Μαργαρέτα. Ακούγοντας ε, τους συναδέρφους, όπου και αν ζούμε, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο θλιβερό είναι να μην μπορούν όλοι να έχουν ε, φωνή επίσης όρης και να μην μπορούν ε, όλοι να ψηφίσουν για να ακουστεί η φωνή τους. Σεσίλια, Κρίμα που δεν το βάλαμε νωρίτερα στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα. Ξέρω ότι εγώ είχα διαφωνήσει, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον αν υπήρχε περιθώριο να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό που είπατε για τη σκοτία είναι ενδιαφέρον. Ότι εκείνοι λένε ότι θέλουν να ψηφίσουν. Όταν κάποιος πληρώνει φόρους πρέπει να έχει λόγο στο πώ θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Οπότε έχει νόημα να πει κανεί ότι μόνο όσοι πληρώνουν φόρους αυτοί πρέπει να αποφασίζουν και για τον τρόπο που δαπανώνται. Αλλά μπορούμε και να το αντιστρέψουμε γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα πολιτικά. Έτσι όπως έχει σήμερα η κατάσταση στις ευρωεκλογέ, για παράδειγμα, όλοι έχουμε δικαίωμα να συμμετέχουμε στις ευρωεκλογέ όπου και αν ζούμε. Και όλες οι χώρες δέχονται ότι μπορεί κανείς να ψηφίσει στις τοπικές εκλογές, ακόμα και αν δεν είναι υπήκος της χώρας δηλαδή. Τώρα, εδώ δεν πρόκειται για φόρους, δεν πρόκειται για εθνικά ζητήματα. Το δημοψήφισμα αυτό έχει να κάνει με το κατά πώς θα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ζωή. Είτε ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν, είτε ζουν αλλού οι πολίτες του, πρέπει να μπορούν να έχουν λόγο. Μήπως θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα για το τι κάνουμε. Στους ε, συμπολίτες μας εξακολουθούν να είναι συμπολίτες μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θλιβερό που δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα, αλλά μη τι άλλο να τους πούμε παραμείνετε μαζί μας για να μπορούμε να έχουμε καλές αποφάσεις. Θα μας λείψετε φοβερά αν τυχόν δεν παραμείνετε μαζί μας. Να είναι αυτό το μήνυμα που θα στείλουμε. Θα έπρεπε να ήμασταν σε θέση να είχαμε μπορέσει να το λύσουμε. Κρίμα. Και βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να είναι πρόθυμο να βρει μια λύση. Αλλά θα του χωρέσουμε αν τελικά το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα είναι να παραμείνουν μαζί μας. Προέδρο. ακούσατε την Μάργαρετέ, ε? πολύ σοφή σε αυτά που είπε. Τώρα, αν θέλετε, Μπορώ να σας ξαναδώσω το λόγο, αλλά πάρα πολύ σύντομα παρακαλώ για να συνοψίσετε και μετά θα προσπαθήσω να καταλήξω σε συμπεράσματα. Οι αναφέρουσες λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο. Για να απαντήσω στην εκπρόσωπο της Επιτροπής. Δεν φτάνει ο έλεγχος. Και το ότι θλίβεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φτάνει. Όπως είπανε και οι Βρετανοί ευρωβουλευτές, και εγώ θα ήθελα στην Ισπανία να ξέρετε ότι στο χωριό μου είναι 30% οι Βρετανοί και δεν έχουμε δικαίωμα. Και αυτά τα δικαιώματα μας αφαιρούνται. Για το δημοψήφισμα, εντάξει, πολύ λίγα μπορούμε να κάνουμε και είναι και πολύ αργά τώρα. Αλλά στραφούμε προς το μέλλον και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να φερούνται τα δικαιώματα ψήφου από τους Ευρωπαίους πολίτες και να μην μπορούν να έχουν λόγο. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να διασφαλίζετε τα δημοκρατικά δικαιώματα σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, η άλλη αναφέρουσα. Να συμπληρώσω και εγώ ότι το δικαίωμα ψήφου είναι τόσο βασικό θεμελιώδες δικαιώματα και αναπόσπαστο από την ίδια την φύση του Ευρωπαίου πολίτη και των δικαιωμάτων του. Οπότε είναι τροπή που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν εμπλέχτηκαν περισσότερο για να διασφαλίσουν ότι αλλάζει ο νόμος του Ηνωμένο Βασίλειο πριν γίνει αυτό το δημοψήφισμα το τόσο σημαντικό. Και σας ζητώ να πάρετε ό,τι μέτρα μπορείτε ώστε να αλλάξει η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επίσης και στις άλλες χώρες μέλη που αναφέρθηκαν σήμερα, ώστε να διορθωθεί αυτή η τεράστια αδικία. Προεδρο. τώρα ευχαριστώ πολύ όλους σας. Τώρα, εκ μέρου τη Επιτροπή μα, θέλω να εκφράσω την ε, απόλυτη κατανόησή μου για την κατάσταση αυτή που αναφέρετε και στην οποία βρίσκεστε. Ως Ευρωπαίοι πολίτες εννοείται ότι έχετε το αδιαφυσβήτητο δικαίωμα ψήφου και αυτό το δικαίωμα σας το έχουν στερήσει. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για το περιεχόμενο της απόφασης που πήραμε σε επιστολή της 25ης Μαΐου. Το υπογράφει η Helen Jones βουλευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προεδρεύει την Επιτροπή Αναφορών εκεί. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω κάπω σύντομα για το περιεχόμενο τη επιστολή αυτή. Λέει λοιπόν ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αλλάξει την εθνική νομοθεσία που έχει να κάνει με τα δικαιώματα ψήφου των Βρετανών πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Δεύτερον, ότι οι αναφέροντες ε, βρετανικής υπηκότητας καλούνται να υποβάλουν αναφορά στην Βρετανική κυβέρνηση το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα των χωρών μελών. Τρίτον, η επιστολή προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στα πλαίσια της ε, συζήτησης στην Επιτροπή Αναφορών θα λέω ότι στηρίζουμε την κυβέρνηση προκειμένου να αλλάξει την νομοθεσία αυτή. Εννοείται ότι το υποστηρίζουμε απόλυτα κι εμείς και ότι θέλουμε να τους ανθαρρύνουμε να αλλάξουν την νομοθεσία. Όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Και συστήνουμε ακριβώς αυτή η πρόταση να πάει από την κυβέρνηση στην Βουλή των Αντιπροσώπων όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εννοείται ότι αφήνουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά μέχρι την δημο την ε, δημοσιοποίηση της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια του 2016, που μεταξύ άλλων θα αναφέρεται και στην αντίφαση αυτή που υπάρχει μεταξύ του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά από την άλλη και τα εμπόδια που υπάρχουν προκειμένου να ασκούν παντού τα δικαιώματά τους. Προτείνω επίσης να υποβάλουμε προφορική ερώτηση, να ενημερώσουμε τους συντονιστές, με ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα λέει πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει συνέχεια στα συμπεράσματα της ανακοίνωσής της του 2014. Αναφέρθηκε και η κυρία Μουσάμερ πριν σε αυτό. Και εσείς το είπατε, το κύριο Τίμερμανς ουσιαστικά δεσμεύτηκε να παρακολουθήσει αυτή την υπόθεση από κοντά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώ έτσι θα προβάλλουμε και πάλι το θέμα μέσω μιας τέτοια προφορικής ερώτηση Και θέλω και να διευρύνω λίγο το πεδίο και θα έλεγα να στείλουμε και επιστολή σε όλες τις χώρες μέλη που έχουν τέτοια στέρηση ε, δικαιώματος ψήφου για τους πολίτες τους. Σε όλες τις μόνιμες αντιπροσωπείες δηλαδή των χωρών αυτών να σταλεί η επιστολή. Συμφωνείτε? Καλώς αυτό και θα κάνουμε. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε από τις χώρες όπου διαμένετε εδώ για να μας μιλήσετε για αυτά τα θέματα. Πολύ σημαντική η συζήτηση γιατί είναι θέμα αρχής. Τι σημαίνει το να είναι κανείς Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό ακριβώς είναι και το ζήτημα που παρακολουθούμε όλοι στενά για τους Βρετανούς. Να ξέρετε πάντως πως όλοι σήμερα νιώθουμε, Ευρωπαίοι, ε, συγγνώμη, Βρετανοί πολίτες. Και περνάμε στο επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη που είναι αναφορά. Έχουμε τέσσερις μάλλον αναφορές μαζί όσον αφορά το βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα και το κλείσιμο βουλγαρικής τράπεζας. Οι αναφέροντες δεν είναι εδώ παρόντες στην αίθουσα. Οπότε θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Έχουμε υποβάλει την απάντησή μας ήδη τον αύριο. Η υπόθεση αυτή αφορά κλείσιμο τράπεζα το 2014. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες τέσσερι ε, βουλγαρικές ε, τράπεζες που βρέθηκε σε ιδιαίτερη δυσκολία και οι καταθέτες δεν μπόρεσαν ε, να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Επέστησαν λοιπόν την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεπώς ξεκίνησε μια διαδικασία επιπαραβάση και απευθύθηκε στις βουλγαρικές αρχές για την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Οι διαδικασίες ε, επί παραβάση έχουν να κάνουν και με την ελεύθερη κυκλοφορία ε, κεφαλαίου. Η βουλγαρική κυβέρνηση τροποποίησε έκτοτε την νομοθεσία και άλλαξε τα πράγματα στο να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους οι καταθέτες και υπήρξε και συντονισμός και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία έστειλε επιστολή στην Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας, που είναι και ο επόπτης σε αυτή την περίπτωση, για να του ζητήσουν ή να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους ή να αποζημιωθούν. Και να ανακληθεί η άδεια για την τράπεζα αυτή, γιατί μόνο τότε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους οι καταθέτες. Πράγμα το οποίο έγινε. Οπότε 100% των καταθετών έχουν πληρωθεί σήμερα σχεδόν. Οπότε έχει κλείσει και η διαδικασία επί Υπάρχει μια νέα οδηγία βέβαια που άρχισε να ισχύει από το 2015. Έχει ενσωματώσει το εθνικό της δίκαιο η Βουλγαρία και αυτήν την οδηγία και εμεί το λέξαμε, λέξαμε την ενσωμάτωση αυτή και ιδιαίτερα για μια ρήτρα που ήταν προβληματική στην προηγούμενη περίπτωση. Δεν είχε ενσωματωθεί σωστά η προηγούμενη οδηγία. Τώρα λοιπόν αυτό έχει γίνει, οπότε πιστεύουμε ότι μπορεί να κλείσει η αναφορά αυτή, εφόσον οι καταθέτες πήραν τα χρήματά τους. Πάρα πολύ μικρά ποσά μένουν ακόμα να διεκπαιρεωθούν, αλλά βασικά το πρόβλημα έχει λυθεί και η Βουλγαρία έχει τροποποιήσει την νομοθεσία της. Ωραία. Ποιος θέλει το λόγο? Κανείς? Η κυρία Κούνεβα. Παρακαλώ κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εξαιρέτηση αναφορά αναφοράς για την ε, Κοπεραντίνα Ταργόφσκα Βάνκα και η παρέμβαση της Κομισιόν αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν ένα θέμα έλθει στην επιφάνεια υπάρχει τρόπος να παρεμβούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί υπέρ του δίκαιου των πολιτών. Η αναφέρον σχετικά με την Κοπορατήνα Ταργόσκα Μπάνκα κάνει μια επισήμανση που πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη εδώ στην Ευρώπη, στην Επιτροπή Αναφορών. Μιλά η εκτεταμένη διαφθορά. Αυτή η εκτεταμένη διαφθορά βάζει πολλά εμπόδια στους βούλγαρους πολίτες, οι οποίοι πολύ συχνά αναγκάζονται να υποκύπτονται σε πολύ σκληρούς τραπεζικούς όρους, να χάνουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους με μεγάλη ευκολία και να βρίσκονται στο έλεος των τραπεζών. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα με μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε τις υποτέσεις που αφορά τα προβλήματα των πολιτών στη Βουλγαρία. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πέτερ. Εγώ έχω να πω το εξή. Το ίδιο το γεγονός ήταν βεβαίως ιδιαίτερα λυπηρό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί ότι ευτυχώ, ευτυχώς στο διάστημα αυτό βρέθηκε μια λύση και γι' αυτό μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Θεωρώ ότι και η διαδικασία της αναφοράς αυτής συνέβαλε με τον τρόπο της στο να δοθεί μια λύση. Συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Πρόκειται για νομικό σφάλμα το οποίο οδήγησε σε δυσμενεί επιπτώσει για του αναφερόμενου. Αλλά από ό,τι κατάλαβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα στο μεταξύ έχει λυθεί. Και ε, εύχομαι να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο ποτέ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου να ζητούν το λόγο. Προτείνω λοιπόν το εξή. Επειδή τα θέματα που περιλαμβάνει η αναφορά φαίνεται να έχουν επιληθεί με επιτυχή τρόπο, ενδεχομένως ίσως και χάρη στις αναφορές σας, ελπίσουμε, οι δράσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ήταν σωστή, η εποπτεία έγινε σωστά, οι διαδικασίες παραβιάσεως έχουν ολοκληρωθεί και η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο τη οδηγία είναι ικανοποιητική. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ συμφωνώ με τον Πέτερ Γιάρ να κλείσουμε τις αναφορές και να προωθήσουμε τις ε, πληροφορίες στου αναφερόμένου. αναφερόμενους. Ευχαριστώ λοιπόν. 2269 είναι η επόμενη ε, αναφορά για το άνοιγμα λογαριασμού, τραπεζικού λογαριασμού σε άλλες χώρες της ΕΕ. Πρόκειται για αναφορά του κ. Μικελάντζελο Ρασπίνα που είναι από σήμερα αλλά παρακολουθεί τη συζήτηση από το διαδίκτυο στην Ιταλία. Και καλά κάνει γιατί εδώ βρέχει συνεχώς. Δίνω το λόγο αμέσως στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια υπόθεση όπου ο αναφέρον ζει στην Ισπανία αλλά επιθυμεί να έχει ε, σύνδεση τηλεφωνική και σύνδεση ίντερνετ στη Γαλλία. Λαμβάνει απάντηση από τον πάροχο της Τελεκόμ ότι έπρεπε να ανοίξει λογαριασμό γαλλικό, σε γαλλική τράπεζα για να μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και ο αναφέρον ε, ε, διερωτήθη αν αυτό ε, παραβιάζει τον κανονισμό ΣΕΠΑ. Η Κομισιόν εξέτασε το θέμα και συμφώνησε με τον αναφέροντα. Πριν να συνεχίσω λοιπόν για τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα ήθελα να εξηγήσω ότι μετά από την μετακίνηση του ε, ΣΕΠΑ, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι σε κάποια αρκετά κρατημέλη οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν ήταν σε θέση να λύσουν ε, το θέμα της μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΣΕΠΑ. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους χρήστες ε, υπηρεσιών πληρωμών, γιατί οι εθνικές αρχές δεν είχαν αρμοδιότητες όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Άρα λοιπόν η Κομισιόν ε, ε, ταυτόχρονα με την παραλαβή της αναφοράς ξεκινήσαμε διαδικασίας, διαδικασία ε, στη Γαλλία για να διερευνήσουμε κατά πόσο οι εθνικές αρμόδιες τους αρχές ήταν σε θέση να λύσουν τη μη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΣΕΠΑ. Λάβαμε στα τέλη του 2015 επιβεβαίωση από τις γαλλικές αρχές πως όντως οι αρμόδιες αρχές τους δηλαδή η Τράπεζα της Γαλλίας και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΣΕΠΑ. Γι' αυτό και στην αναφορά ε, συμβουλέψαμε τον αναφέροντα να στείλει αυτή την υπόθεση και όλα τα σχετικά στοιχεία σε τις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας. Του προτείναμε μάλιστα να τα στείλει και στην Κομισιόν αν ήθελε, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση του. Συνάδελφοι, Πίτερ, θες το λόγο? Πέτερ Γιάρ. Με την πρώτη ανάγνωση λέει κανείς, μα δεν είναι δυνατόν διότι ε, η ιδεολόγηση έχει γίνει με την βάση τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Μετά ε, ακολούθησε νέα διαδικασία. Μπορεί λοιπόν τώρα να μεταφέρει κανείς χρήματα χωρίς πρόβλημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι αυτό που γίνεται εδώ και που καταγγέλλεται είναι παράνομο στην ουσία. Και οι εθνικές αρχές δεν έχουν κάνει τίποτε για να το σταματήσουν. Μιλούμε για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάποια αναπτυσσόμενη χώρα. Νομίζω ότι η ε, Κομισιόν έχει δίκιο. Νομίζω πάντως ότι εάν θέλουν οι εθνικές αρχές μπορούν κάτι να κάνουν. Μπορεί να επιβληθεί και πρόστιμο στην ε, επιχείρηση που κάνει αυτά τα πράγματα, εφόσον πρόκειται καθαρά για παραβίαση των κανόνων της ενιαίας αγοράς και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και ακριβώς γι' αυτό υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, για να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πρώτον, να μην λοιπόν η αναφορά ανοιχτή. Δεύτερο, να επιληφθεί και η Επιτροπή μας που ασχολείται με την ενιαία αγορά. Να τους διαβιβάσουμε την αναφορά, να δουν δηλαδή τι πράγματα γίνονται. Τέλος, πρόκειται για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Να ενημερωθεί λοιπόν αναφερόμενος, να ε, ενημερωθούν και οι γαλλικές αρχές, διότι πρόκειται καθαρά για παράνομη ε, δραστηριότητα. Μάλιστα και μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη θέση σου, Πίτερ, ότι αυτή η οδηγία 260 του 2012 είναι η ισχύουσα νομοθεσία για τις ενιαίες ευρωπαϊκές πληρωμές. Είναι κανονισμός και πρέπει να ακολουθείται και να εφαρμοστεί παντού. Πλήρως. Η Γαλλία λοιπόν επιβεβαίωσε ότι υιοθέτησε μέτρα για να εξασφαλίσει την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, ιδιαίτερα το άρθρο 9, αλλά χρειάζεται η Κομισιόν να συνεχίσει να παρακολουθεί τι γίνεται και άρα να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, αλλά να ενημερώσουμε και τον αναφέροντα ότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και ότι η Κομισιόν έχει τώρα το αίτημα λάβει από την Επιτροπή μας να ερευνήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται στους πελάτες ε, να έχουν λογαριασμό σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Πρόκειται λοιπόν για σαφή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η απέτηση για γαλλικό λογαριασμό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και ο αναφέρον θα πρέπει να ενημερωθεί ότι αυτή είναι η ερμηνεία μας και ότι τώρα η Κομισιόν το εξετάζει και θα επανέλθει αργότερα. Έτσι λοιπόν κλείνουμε αυτό το θέμα, μάλιστα. Εγώ θέλω να διαβιβαστεί στην ε, Επιτροπή Ενίας Αγοράς να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αυτή η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να επιληφθεί και αυτή του θέματος. Παρακαλώ επίσης την Κομισιόν στην επιστολή που θα αποστείλει στις εθνικές αρχές, κατά πάσα πιθανότητα, να δείξει και την ανυπομονησία της. Δεν είναι δυνατόν να μην επιλύεται ένα τέτοιο πρόβλημα. Εάν θέλουν οι εθνικές αρχές δηλαδή αν θέλουν, μπορούν να το ξεκαθαρίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το καταλαβαίνω. Η υπόθεση είναι γνωστή. Δεν είναι δυνατόν οι εθνικές αρχές να παρασταίνουν σαν να μην ξέρουν τίποτε. Ευχαριστώ. Ασφαλώς θα στείλουμε την ε, αναφορά στην ΙΜΚΟ για ενημέρωση αλλά και για να εμπνευστούν να αντιδράσουν. Ε, μου φαίνεται ότι το διάλειμμα για το μεσημεριανό θα είναι κάπως ε, μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως. Σας ξαναδώ λοιπόν το απόγευμα στις 3.